Έχουμε ένα σχέδιο έκθεση, έκθεσης για την ε, εκπροσώπηση των εργαζομένων στα δουσού των εταιριών στην Ευρώπη. Ο Ενρίκο Γκάσπαρα είναι ο εισηγητής. Έχετε το λόγο, αγαπητέ συναδελφέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους που υπέβαλαν 60 τροπολογίες, πολύ ενδιαφέρουσες, μπορούν να συνεισφέρουν στο να βελτιωθεί η πρόταση νομοδότησης που έχω Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι η πρόταση γνωμοδότησης που έχω υποβάλει έχει σαν νομική βάση το άρθρο 143 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στο να εκφράσει μία νομική άποψη, ελπίζω σοβαρή, ε, ενιαία, όσο πιο ενιαία γίνεται. Βεβαίω υπάρχουν κάποιε αποκλήσει σε διάφορε τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τι επεξεργαστούμε, ούτω ώστε αυτή η απόκληση που παρατηρούμε να καλυφθεί, α πούμε, να υπάρξει μια απόπειρα σύγκληση. Θέλουμε να εναρμονίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο την ισχύουσα νομοθεσία. Σε σχέση με τις 18 χώρες που έχουν ήδη εφαρμόσει την νομοθεσία, ε, η απόπειρα είναι να υπάρξει εναρμόνιση και των 28 χωρών. Να μην πλήξουμε την αυτονομία των κρατών βεβαίως, ε, γιατί εδώ εφαρμόσουμε την αρχή της επικουρικότητας και θέλουμε σίγουρα να τη σεβαστούμε αυτή την αρχή. Σας ευχαριστώ όλους. Ελπίζω ότι και στη σημερινή συζήτηση και στην επόμενη συζήτηση που θα έχουμε τους σκιώδεις ε, εισηγητές στις 10 Μαΐου στο Στρασβούργο, αλλά και σε αυτή που είχαμε στο παρελθόν με τους σκιώδεις εισηγητές, να μπορέσουμε εν ευθέτω χρόνο πριν από την ε, συνεδρίαση ήδη της 10ης Μαΐου να κάνω μια πρόταση στους συναδέλφους, συμβαστική πρόταση, που ελπίζω ότι θα εξασφαλίσει ευρεία συνένεση. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και ευχαριστώ κυρίως αυτούς που συνεισέφεραν στη δουλειά μας, στο κείμενό μας. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την παρουσίαση. Ευχαριστώ για το ανοιχτό του πνεύμα, τη διαθέσιμότητά του να συνεργαστεί με τους κοιόδης εισηγητέ για το κείμενο αυτό, που σκοπό έχει να εξασφαλίσει εκεί όπου το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία, οι εργαζόμενοι να εκπροσωπούνται στα διοικητικά συμβούλια, ούτω ώστε με συνεχεία τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν το πώς θα εκπροσωπηθούν ε, και το αν θα έχουν ε, δικαίωμα ψήφου. Με σεβασμό της ε, επικουρικότητας και με σεβασμό της αρχής ότι οι ίδιες εταιρείε αποφασίζουν για τα οργανωτικά τους θέματα, τα εσωτερικά οργανωτικά τους θέματα. Να δείξω κάποια θέματα τώρα σε ό,τι αφορά την τροπολογία 20. Θα πρέπει το προσωπικό της Επιτροπής να δει αν αυτή η τροπολογία έγινε προκειμένου να αποσυρθεί η οδηγία και αν συνάδει με τους νομοθετικούς κανόνες. Γιατί εμείς προτείνουμε κάτι στην Κομισιόν. Μα αυτό δεν είναι ένα έγγραφο τέτοιου τύπου. Πιστεύω ότι θα βρούμε μια καλή ισορροπία πάντως, ούτω ώστε να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο για τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να εκπροσωπηθούν εργαζόμενοι. Δεν θέλω όμως να αρχίσω μια άλλη συζήτηση. Θέλω να ρωτήσω αυτούς που ξέρουν τα θέματα αυτά, να μου πούν ποια είναι η καλύτερη δομή για την εκπροσώπηση των εργαζομένων. Όταν μιλάμε για εργαζόμενους, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν μια συμβατική σχέση εργασίας. Μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν νόμιμα. Δεν μιλάμε φυσικά για τη μαύρη αγορά. Τι εκπροσώπηση θα μιλήσουμε εκεί για αυτούς τους εργαζόμενους. Ε, thank Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρέγκνερ, πολύ σύντομα. Για τα επιχείρηματα που προβάλλατε εσείς είναι ζήτημα που έχει να κάνει και πρέπει να διευκρινιστεί, το έχουμε εκκρεμές εδώ και κανένα δύο χρόνια, πρέπει ίσως να καταλήξουμε πια σε μια απόφαση στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι με αφορά ιδιαίτερος και επί τη ευκαιρία θα ήταν σκόπιμο με τον εισηγητή κύριο Τεγκράντε Πασκουάλ να συζητήσω ποια είναι η δική του θέση και ίσως διμερώς μπορούμε να το λύσουμε κατά τα άλλα. Θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερος ευχαριστώ τον κύριο Κασπάρα για την πολύ καλή δουλειά του, για τι ε, τροπολογίε του, μία κυρίω που έχω καταθέσει, το δικαίωμα για ενημέρωση και συμμετοχή στις συνομιλίε είναι θεμελιώδε δικαίωμα δεν πρέπει ε, να αφήσουμε να μας ξεφύγει αυτό ως δικαίωμα. Καταγράφεται και στον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει μέσα από την εκθέση αυτή απλώς να διευκρινιστούν οι όροι λειτουργίας του. Και επίσης υπάρχει μια άλλη τροπολογία που έχω καταθέσει εγώ. Ο υπεύθυνο για τη συν απόφαση, συν διαμόρφωση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το σύστημα συναπόφαση μπορεί να ισχύει εκεί. Πρόκειται για ένα ε, εργαλείο σημαντικό ανάλογα με το μέγεθος επιχείρησης, μεγάλη, πολύ μεγάλη, μέτριου μεγέθους και έχει πολύ ενδιαφέρον να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα. Ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω να ζητεί κανείς άλλο το λόγο. Θέλει ο κ. Γκάσπαρα να σχολιάσει. Να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά του συναδελφούς. Όπως είπε και στην εναρκτήρια παρέμβασή μου, νομίζω ότι ήταν σημαντική η παρέμβασή τους, δηλαδή οι 60 τροπολογίες που υπέβαλαν και εγώ θα προσπαθήσω να βρω συμβιβαστικές λύσεις, ούτως ώστε να είναι συνενετική αυτή η έκθεση και ή άλλω στην έκθεση Handel θα ε, υπάρχει δυνατότητα η Επιτροπή να μπει σε, στην ουσία του θέματο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν το 9 και πάμε στο 10. Εξέταση τροπολογιών. σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Α, όχι, δεν είναι εδώ οι εισηγητές. Η συγγετρία κυρία Χάουταλα. Να περιμένουμε μερικά λεπτά ίσως για να ενημερωθούμε αν ε, έρχεται. Uh, uh, λοιπόν, δεν έχουμε εισηγητή, την εισηγητρία για τα επόμενα λεπτά. Γι' αυτό προτείνω να κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 4 και 10. 4 και 10. όπου θα δούμε το 10 της κυρίας Χάουταλα και μετά τον Επίτροπο Χίλ, αν δεν έχετε αντίρρηση. Διάλειμμα λοιπόν μέχρι τι και 10.